αλλά θα παραμείνουν αρκετά χαμηλότερες, χαμηλότερα ε, από, τις 100, 133 ευρώ των ΗΠΑ ε, και τα, τα 130 ευρώ της Κίνας. Είμαστε αρκετά φθηνότεροι στην Ευρώπη σε αυτό το θέμα. Επίσης συμφωνήσαμε το Συμβούλιο για θέματα για το θέμα που είναι πολύ λεπτό περί της σύνδεσης ε, της, της, παραχώρησης της έκδοσης θεωρήσεων ε, και της αποδοχής της επιστροφής ε, αυτών που έχουν εισέλθει παράνομα στις χώρες τους, του, της Ζων Σέγγεν. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ, ε, για την προσήλωσή του. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τον κύριο Μπέκερ και την κυρία Βερζιά ε, για την πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ για τους ε, συνεργάτες μας. Και τελειώνω, πρώτα. 30 χρόνια είμαι ευρωβουλευτής. Και αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση. Ένα έχω να πω. Το πιο όμορφο πολιτικό σχέδιο είναι η υλοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος. Ζήτω η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, γινόμαστε όλο και πιο συναισθηματικοί. Και περιμένετε να ακούσετε τις δικές μου καταληκτικές παρατηρήσεις. Η κυρία Βερζιά, ε, 1,5 λεπτό. Ε, οι μετακινήσεις πληθυσμών είναι πιο σημαντικέ από ό,τι ποτέ στον κόσμο. Ένα δισεκατομμύριο άτομα μετακινούνται κάθε χρόνο από μία χώρα σε άλλη, ιδιαίτερα στο βορρά. Κύριε Ντεπρέ, 500 εκατομμύρια άτομα έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. 250 ε, εκατομμύρια άτομα είναι μετανάστες. Δηλαδή παραμένουν πάνω από ένα έτος σε, κάποιο, σε κάποια χώρα. Για διάφορους λόγους μεταναστεύουν. Ε, Παρόλε τι προσπάθειε του εισηγητή, όμω ο κώδικα αυτό δεν είναι ισορροπημένο. Δεν ισορροπεί ανάμεσα στη διευκόλυνση των τουριστικών ε, ταξιδιών, ε, την, νο, παράτυπη και την νόμιμη μετανάστευση. Παρόλες της πραγμα... την πραγματικότητα, παρόλου τους θανάτους, ε, εστιαζόμαστε όλο και πιο πολύ στον έλεγχο των συνόρων και στην διαχείριση ε, της παράτυπης μετανάστευσης. η η νόμιμη μετανάστευση όμως είναι 20 φορές πιο σημαντική σε νούμερο από ό,τι η παράτυπη. 2,5 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο. Η πραγματικότητα είναι ότι ε, κλείνουμε την πόρτα τελικά στους πρόσφυγες ε, και ε, με λυπεί τις δύο τελευταίες θητείες που ήμουν εδώ, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη έχουν αρνηθεί να δημιουργηθούν ανθρωπιστικές θεωρήσεις. 90% των ατόμων στα στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση δίδει διεθνή προστασία τα τελευταία τρία χρόνια έχουν φτάσει με παράτυπο τρόπο. Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερη στην απόδοσή μα. Επειδή είναι δική μου τελευταία παρέμβαση, θα ήθελα και εγώ λίγο παραπάνω χρόνο, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλου όσοι με έχουν βοηθήσει τι τελευταίε δύο Βλέπω πολλού συναδέλφου με του οποίου με πολύ χαρά συνεργάστηκα ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, το προσωπικό μας, τα στελέχη μας, τους συνεργάτες μου, αλλά και όλους τους υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορατούς και αόρατους, τους διερμηνείς, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε σε εξαιρετικές συνθήκες, άνθρωποι τους οποίους δεν βλέπουμε συχνά, παρόλα αυτά είναι παρόντες. Πολύ, πολλά ευχαριστήρια. Θα συνεχίσω να παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον και προσοχή το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι ένα άχρηστο όργανο όπως νομίζουν κάποιοι πολίτες, συμπολίτες μας ε, εξαιτία λαθασμένων προσεγγίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί τα επιτρέπω αυτά, για έναν πολύ ρεαλιστικό λόγο. Ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο ε, θα έχουμε όλους τους συναδέλφους όταν λέω τα ίδια πράγματα να χειροκροτούν. Βάλερο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Για να δω, αν και εγώ θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχω. Κώδικας θεωρήσεων. Ήταν ο πρώτος φάκελος που είχα πάρει από την πολιτική μου ομάδα τους πράσινους και είναι η τελευταία μου παρέμβαση για το ίδιο θέμα σήμερα στη θητεία. Στο ξεκίνημα της θητείας μας είχαμε ξεκινήσει με μια πολύ καλή πρόταση από την Επιτροπή η οποία προσπαθούσε να διευκολύνει την κατάσταση για πολλούς ανθρώπους που ήθελαν να έρθουν στην Ευρώπη ε, και διευκολυνόταν το ενδεχόμενο να έρχονται περισσότερες φορές. Βέβαια η πρόταση αυτή μπλόκαρε στο Συμβούλιο, δεν ήθελε να συμφωνήσει με τη δική μας πρόταση μεταξύ άλλων για την ανθρωπιστική θεώρηση. Μετά πήραμε μια νέα πρόταση που ήταν τελείως διαφορετική, καθόλου κοντά στην αρχική, δεν είχε στόχο να διευκολύνει, αλλά να ασχολείται κυρίως με την σύνδεση των θεωρήσεων με την επιστροφή των ατόμων. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να βελτιώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου στο κείμενο αυτό, ωστόσο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και πάλι όλα όσα θέλαμε να πετύχουμε. Η σύνδεση με τις επιστροφές στο κείμενο αυτό είναι ο λόγος για τους οποίους εμείς οι πράσινοι δεν θα υπερψηφίσουμε την έκθεση παθότι έχει πολλά θετικά στοιχεία. Τα τέλη. Τα τέλη θα αυξηθούν. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο για επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, για οικογένειες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη από φτωχέ χώρες να πληρώνουν τέτοια τέλη θεώρηση. Θα είναι δύσκολο τα άτομα αυτά να πληρώσουν το ποσό αυτό. Βλέπω, πρόεδρο, ότι αρχίζετε και κουνάτε τα χέρια σας. Κλείνω ευχαριστώντας όλους σας για την εξαιρετική συνεργασία και ό,τι καλύτερα σε όσους ε, θα ξανάρθετε και σε όσους φύγουν. Ευχαριστώ κύριε Βαλέρο. Ο κύριος Άκερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ο ορισμός του κράτους είναι πολιτική οντότητα με μονοπόλιο του ελέγχου στα εξωτερικά της σύνορα. Οι θεωρήσεις είναι ένα άλλο παράδειγμα όπου η Ευρώπη προσπαθεί να περάσει για κράτος. Το κάνει όταν νομοθετεί για την ε, αλληλεία ξεκίνησε, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας το έκανε και, στους διεθνείς, ε, και στις διεθνείς σχέσεις. Και τώρα έρχεται στον κώδικα θεωρήσεων άλλο η εναρμόνιση. Εδώ η εναρμόνιση στην ουσία έχετε σε αντίθεση με την ε, επικουρικότητα. Η Ένωση δεν μπορεί να πάρει κάτι τέτοιο και εμείς αυτό στη Βρετανία δεν το δεχόμαστε. Οι απαιτήσει θεώρηση είναι αρμοδιότητα των κρατών, όχι της Ένωσης. Επιτρέπουμε σε τρίτες χώρες να στείλουν ε, κόσμο εδώ, αλλά αυτό, ιδίω η προσπάθεια να ε, συνδέσουμε την ε, επιστροφή με τις θεωρήσεις είναι βασική αρχή της εθνικής, του, της εθνικής κυριαρχίας. Προχωρώντας προς την κατεύθυνση αυτή θα αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Δεμπρετών, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλλαγή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Θεωρήσεων που εξετάζουμε σήμερα έχει επίσημα ως στόχο να διευκολύνει, παραθέτω, το ταξίδι πολιτών τρίτων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται λοιπόν για νέο εργαλείο μετανάστευση το, με το οποίο αντιτίθεμε αποφασιστικά. Η κτήση θεωρήσεων ε, βραχίας διαμονής διευκολύνεται με άφρονα τρόπο. Κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των κινδύνων ε, κατάχρησης, ιδίως όταν ε, τα αιτήματα υποβάλλονται στα σύνορα. Η άρνηση έκδοσης θεωρήσεων σε πολίτες ε, της τρίτου, τρίτων χωρών που αρνούνται να πάρουν πίσω τους πολίτες τους είναι ένα καλό μέτρο το οποίο ωστόσο παραμερίζεται. Οι συνθήκες υλοποίησης δε αυτής της διαδικασίας είναι τόσο σύνθετες που δεν δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στη διάταξη αυτή. Το κείμενο προέβλεπε αρχικά να υπάρξει ένα νέο δίκτυο νόμιμης μετανάστευσης με ένα ευρωπαϊκό ανθρωπιστικό, με μια ε, ευρωπαϊκή ανθρωπιστική θεώρηση που δεν, ήταν και, που δεν κατάφερε ούτε καν να μειώσει την παράνομη μετανάστευση. Ευτυχώς αυτή η παράλογη ιδέα ε, καταργήθηκε. Έχουμε μπροστά μας μια μαζική ε, μετανάστευση που σχετίζεται με τις δημογραφικές εξελίξεις θα έχουμε, το ότι θα έχουμε λίγες χιλιάδες νόμιους μετανάστες δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια παράνομων. Το σύστημα Σέγγεν έχει, έχει καταρρεύσει, έχει αποτύχει. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η τελευταία παρέμβασή μου σε αυτή την ε, θητεία μου θυμίζει μου επιτρέπει να θυμίσω στο Κοινοβούλιο την, ε, τα σημαντικά. Η πραγματική συζήτηση δεν είναι τα δευτερεύοντα, αλλά το ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του, του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δίας μέρα. 1,5 λεπτό. Θέλω να συγχαρώ τον Χωα Φερνάντο. Ε, ένα το κοινό σύστημα θεωρήσεων είναι σημαντικό όχι μόνο σε θέματα ασφάλειας και πρόληψης παράτυπης μετανάστευσης, αλλά είναι θεμελιώδες για την καλή λειτουργία πολλών οικονομικών κλάδων. Τον τουρισμό, για παράδειγμα. Ο τουρισμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για πολλές περιοχές Ευρώπης. Το 2017 μόνο 14 εκατομμύρια θεωρήσεις Σέγγεν δόθηκαν για βραχυχρόνιες διαμονές. Ε, διαδικασίες ε, πιο ευέλικτες όπως οι ηλεκτρονικές αιτήσει με, ε, με ένα μια έξι μηνών για τις αιτήσει, οι δυνατότητες πολλαπλών θεωρήσεων μακρόχρονη διάρκεια η βελτίωση στη συνεργασία σε θέματα επανεισδοχής είναι ορισμένες από τις βελτιώσεις της πολιτικής θεωρήσεων η αλλαγές αυτές θα βοηθήσουν το εμπόριο, τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και μειώνοντας τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης. Είναι πολύ σημαντικό βελτιώσεις στην πολιτική των θεωρήσεων να γίνονται σύμφωνα ε, με τις προδιαγραφές του CIS και του VIS προκειμένου να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των ε, συστημάτων πληροφοριών. Και εγώ φεύγω, Πρόεδρε. 35 χρόνια δημόσιας ζωής. Μπορώ να, τις, να τα συνοψίσω με μία λέξη. Ευχαριστώ. Ή με δύο λέξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ή στο επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ. Εκ βάθους καρδίας. Φαίνεται ότι αυτή η με δυο λεξεις ευχαριστω πολυ ειστε επανειδην ευχαριστω πολυ εκ μία συζήτηση για τους παρελθόντες. Κλοντ, έχετε το λόγο, κύριος Μουράης. για δύο λεπτά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη ευαισθησία που δείχνετε στην Προεδρία εδώ σήμερα. Το θέμα δεν είναι τόσο πολύ ο κώδικα θεωρήσεων, πιο πολύ είναι ένα αντίο από πολλού συναδέλφου. Αλλά να ευχαριστήσω ό,τι αφορά του θεωρήσει ε, τον εισηγητή για την φιλόδοξη αυτή αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό τη ε, βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων. Όπω είπαν πολλοί συνάδελφοι, θα ήθελα επίση να κάνω και αυτό που έκαναν ε, και οι άλλοι συνάδελφοι με την ευγενική ε, σας, ε, ε, αν μου το επιτρέπετε, είναι η τελευταία συνεδρίαση. Πρόσεξα ότι έχουμε πολλούς συναδέλφους εδώ από την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ και θα ήθελα να πω και προς τον κύριο Μέρα το εξή. Αν ε, διαβάσατε τον κατάλογο των ψηφοφοριών θα δείτε ότι έχουμε απανοτές διαδοχικές εκθέσεις από την Επιτροπή μας. Έχουμε εδώ πολλούς συναδέλφους ε, εμπειρογνώμονες για το Δουβλίνο, τα σύνορα, τις βίζες, ε, το Σέγγεν, το πακέτο ασύλου. Θα δείτε ότι πολλές ήταν οι εκθέσεις που ψηφίστηκαν, πολλές ε, εκθέσεις, Επίτροπε, και αν κοιτάξετε τον επιτροπέ που θα ότι πολλές από τις εκθέσεις μας είναι, έχουν μπλοκαριστεί γιατί έχουμε κάποια από τα πια δύσκολα θέματα. Γιατί είναι και δύσκολο και βαρύ το πολιτικό κλίμα, άλλωστε. Να ευχαριστήσω εκ βάθου καρδίας όλα τα μέλη τη επιτροπή, ΛΥΜΠΕ, με τα οποία είχα το πλεονέκτημα και το προνόμιο να συνεργαστώ. Ποιοτική ήταν η νομοθεσία η οποία παρήγαμε και η μεγάλη μου ελπίδα είναι στην επόμενη θετία να ξεμπλοκαριστούν να ξεπαγώσουν αυτά τα νομοθετήματα, να καταλάβει το Συμβούλιο τι ποιότητα ε, νομοθεσία ε, παρήγα για το Κοινοβούλιο και να καταλάβουν ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι κλωστοσκούφι, είναι ένα όργανο με πολύ ποιοτικού πολιτικούς που παράγουν ε, νομοθεσία υψηλού επίπεδου και ποτέ δεν θα ξεχάσω την εμπειρία αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Mr. Jurek. Ο κύριος Γιούρεκ για ένα λεπτό. Αν δεν φύγετε. Αν δεν να φύγετε, δεν πάρτε και λίγο παραπάνω από ένα λεπτό. Αλήθεια σας λέω. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πέντε χρόνια ήμουν στο Κοινοβούλιο. Υπηρέτησα τη χώρα μου, υπηρέτησα την συνεργασία μεταξύ των εθνών της Ευρώπης και είναι συμβολικό το ότι στο τέλος της θητείας μας συζητούμε για τα σύνορα. Τα σύνορα είναι η ουσία του κράτους. Δεν μπορείς να ανοίξεις. Ε, ε προφανώς είναι καλό να είναι ανοιχτά σύνορα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτόμαστε τους ελέγχους, την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, που εν τέλει θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς έχουμε εργαστεί για τον κώδικα θεωρήσεων και έχω την εντύπωση ότι κάποιες έννοιες ε, δεν έχουν γίνει ε, σαφείς. Υπάρχει μια μακρά συζήτηση για το νόμιμος παράνομος, ή ε, παράτυπος, αλλά σε ένα δεν μπορείς να μιλήσεις για άσκηση κράτους, εφαρμογή κράτους δικαίου όταν μιλάς για παράτυπη είσοδο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε ως έθνη κράτη την, ε, τα σύνορά μας. Η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά που έκανε για τον κώδικα θεωρήσεων. Εκτιμώ την αφοσίωση και αποφασιστικότητα που έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη σημαντική νομική διαδικασία. Υποστηρίζω τι συμβαστικέ ε, λύσει όπου πετύχαμε ε, συμφωνία για τις θεωρήσεις, την θεώρηση πολλαπλών εισόδων ή την θεώρηση ε, μακροχρόνιας διαμονής. Οι ευκαιρίες αυτές θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, να παρακολουθούμε τους κινδύνους ασφάλεια. Συνάδελφοι, είναι η τελευταία παρέμβασή μου στην Ολομέλεια και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους σας για τις εξαιρετικές συζητήσεις που είχαμε, τη μεγάλη, τα την επιτυχία σε πολλά ζητήματα. Δέκα χρόνια υπηρέτησα την ευρωπαϊκή δημοκρατία μαζί με εσά και κάποια στιγμή η πολιτική σταματά, η φιλία ωστόσο παραμένει. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους σας ό,τι καλύτερο στο μέλλον, είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε σε ένα νέο δρόμο στη ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ. Άντερσον, ένα λεπτό. Δυστυχώς αυτή πρόταση είναι μία ακόμα επίθεση στα δικαιώματα και την ασφάλεια των μεταναστών και των τροτών ατόμων. Πολλοί από τους ε, λεγόμενους ε, ε προοδευτικούς υπέκυψαν στις πιέσεις της δεξιάς βάζοντας, ε, προτεραιότητα στην ε, προάσπιση των εξωτερικών συνόρων προκειμένου να κρατηθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή όμως πλούσιοι πολίτε τρίτων χωρών μπορούν να αγοράσουν χρυσές θεωρήσεις ενώ οι στρατιωτικέ παρεμβάσει δημιουργούν πρόσφυγε που δεν έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστικέ θεωρήσεις. Ακόμα χειρότερα, οι πρόσφυγε ανταλλάσσονται με τρίτε χώρε ε, πολλές από τις οποίες έχουν πολύ κακό παρελθόν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σαν να ήταν αυτοί οι άνθρωποι ανεπιθύμητοι, ανεπιθύμητο, ανεπιθύμητα προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει υποχρεώσει να, να βοηθάει όλους και τους πιο ευάλωτους ανεξάρτητα του οικονομικού, της οικονομικής τους κατάστασης. Κανένα άτομο, κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος. Κοράω, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο τουρισμός είναι σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Το 2018 πάνω από 700 δις ευρώ έδωσε στην Ευρώπη και σε 2 εκατομμύρια, ε, 12 εκατομμύρια άτομα σε 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις ασχολούνται με τον τουρισμό. Το 2018 ο κλάδος συνέβαλε στο 3,9% της, του ΑΕΠ της Ένωσης. 5% του εργατικού δυναμικού. Η, άνυ, άνοδος της, ε, ε, του τουρισμού έχει σημαντικές συνέπειες λοιπόν για την Ευρώπη. Η μεταρρύθμιση παρέχει ένα καλό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό επιτρέποντας την διευκόλυνση των θεωρήσεων. Έχω εμπιστοσύνη στο ότι αυτή η νέα μεταρρύθμιση διευκολύνει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες επιτρέποντας την επιστροφή των πολιτών των χωρών αυτών σε κατάσταση ε, πα, παράτυπης παρουσίας. Ε, ταυτόχρονα θα ενισχύσει τις προσπάθειες συνεργασίας με τις χώρες αυτές για τους επαναπτυσμούς. Ο κύριος Κοέλιο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αναθεώρηση του κώδικα θεωρήσεων είναι ακόμα στοιχείο της αναθεωρήσης της πολιτικής της Ευρώπης για τις θεωρήσεις. Με αυτή την αναθεώρηση προσπαθούμε να προωθήσουμε τον τουρισμό, πολύ σημαντικό οικονομικό κλάδο για την Ευρώπη και για την ε, Πορτογαλία και να ενισχύσουμε την ασφάλεια με τις συμφωνίες επανεισδοχής. Θέλουμε να ενισχύσουμε λοιπόν τον τουρισμό βραχύνοντας τις προθεσμίες, διευκολύνοντας τους τουρίστες ε, και κάνοντας πιο ευέλικτες διαδικασίες. Πάρα πολύ σημαντικό σημαντικός ο τομέας κρουαζιέρας, ε, ιδιαίτερα για νησιωτικές περιοχές όπως οι Αζόρες και η Μαδέρα, ε, καθώς επίσης είναι σημαντικές και πολλαπλές θεωρήσεις. Ε, θα διαθέτουμε επίση περισσότερε πληροφορίε, θα συλλέγουμε περισσότερε πληροφορίε και θα κάνουμε περισσότερου ελέγχου και διασταυρώσει πριν την έκδοση των θεωρήσεων. Η επανεισδοχή, από την άλλη μεριά, θα ε, θα, είναι, θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο ώστε να δώσουμε περισσότερη βοήθεια στις χώρες που συνεργάζονται περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό το νομοθέτημα βοηθάει ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνω συγχαρητήρια στον Κλοντ Μωράης και στον κύριο Λόπες. Κυρία Κέγγε, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω Δύο λόγια για την Επιτροπή στην οποία δούλεψα, ως τελευταία παρέμβαση για την Επιτροπή Λίμπε στη θητεία αυτή. Πολλά κάναμε κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. συμβάλαμε στο να υπάρχει ένα, κοινο, ένα ενωσιακό σύστημα ασύλου, ομαδικά. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις διαφορές μας όπου ήταν δυνατό και να στηρίξουμε τις, το έργο μας αξίες μας Όλα αυτά έγιναν ελπίζοντας να βελτιώσουμε την κατάσταση προς όφελος μιας πιο δίκαιης ε, κοινωνίας και ελπίζω η ψήφος των πολιτών να με, να με βοηθήσουν να, επανέλθω. Εδώ, μετά από τέσσερα χρόνια έντονων ε, διαπραγματεύσεων μπορούμε να πούμε με περηφάνεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά μια κοινή πολιτική θεωρήσεων. Και με αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή στην οποία ε, εργάστηκα, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Μία πολιτική που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα και που παραμένει ένα ουσιαστικό εργαλείο για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις είτε για οικονομικούς είτε για ε, τουριστικούς λόγους. Μια πολιτική που θα στρέφεται προς την ανάπτυξη και θα είναι συνεκτική με άλλες πολιτικές της Ένωσης, εμπορικές, ε, πολιτιστικές, ε, τουριστικές. Διευκολύνουμε τις διαδικασίες, μειώνουμε το κόστος και εντοπίζουμε με ακρίβεια το αρμόδιο κράτος μέλος για να εξετάσει μια αίτηση θεώρησης, ιδίως όταν κάποιος θέλει να επισκεφθει πολλα πολλά κράτη-μέλη. Δώστε μου κάποια λεπτά ακόμα, Πρόεδρε, γιατί το πρώτο μέρος της ομιλίας μου ήταν ευχαριστήρες προς την Επιτροπή. Προβλέψαμε τη δυνατότητα να υποβάλουν online αιτήσει οι ετούντε και να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική υπογραφή. Ιδίω διαφυλάξαμε τη δυνατότητα προσφυγή στους ετούντε, στους οποίους οι οποίοι δεν έλαβαν θεώρηση. Τέσσερα χρόνια μακρών διαπραγματεύσεων που επέτρεψαν ωστόσο η μεταρρύθμιση αυτή να παραμείνει στο εσωτερικό ενός ε, θεσμικού νομικού πλαισίου με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο μας βρίσκεται ακόμα με τη συζήτηση, στη συζήτηση αυτή είναι ότι είναι η τελευταία συνδρίαση για πολλούς από τους συναδέλφους μας αυτή. Και έτσι έγιναν και κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις ε, στις ομιλίες για το θέμα της σημερινής διάταξης. Σας ζητώ να δείξετε κατανόηση. Έχουμε τώρα την διαδικασία Catch the Eye και έχουμε τέσσερις συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και μετά θα ζητήσω από τον Επίτροπο τον κύριο Κανιέτε και από τον εισηγητή τον κύριο Αγγίλαρ να πάρουν το λόγο για να ολοκληρώσουν τη συζήτησή μας αυτή. Έχουμε λοιπόν τέσσερις συναδέλφους για το Catch the Eye και άλλες δύο παρεμβάσεις στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σόντροβα έχει το λόγο. Ε, <clears throat> ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κατανοώ 100% το γεγονός ότι είναι η τελευταία, προτελευταία ημέρα της θητείας και δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι όσο συνήθως. Ωστόσο, συζητάμε τον κώδικα θεωρήσεων. Πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω το νέο αυτό κώδικα θεωρήσεων και πιστεύω ότι ο συμβιβασμός είναι καλός. Απλοποιεί τη διαδικασία για όσους ε, ταξιδεύουν νόμιμα και είναι καταχωρισμένοι στο σύστημα, οι οποίοι δεν χρειάζεται πλέον να έχουν φυσική παρουσία για την υποβολή του αιτήματο για τη χορήγηση θεωρήσεων. Επίση, σε ό,τι αφορά τη μακρά διάρκεια των πολλαπλών θεωρήσεων, θεωρήσεων πολλαπλή ε, εισόδου. Από την άλλη, ενισχύουμε και την ασφάλεια. Και αυτό είναι σημαντική πτυχή σε ό,τι αφορά και την ε, απειλή τη μετανάστευση εδώ οι κανόνες καθίστανται πιο αυστηροί. Και έχουμε και διάφορα μέτρα για τις επιστροφές. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Συζητούμε τον κώδικα θεωρήσεων που είναι βεβαίως μια σημαντική διαδικασία γιατί αποσκοπεί στο να βάλει τάξη στο ποιοι μπορούν να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή όμως κύριε Πρόεδρε συνεχίζεται η διαδικασία καραντίνας απέναντι σε όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο από την Αθήνα στις Βρυξέλλες με παράνομους ελέγχους διαβατηρίων στο αεροδρόμιο Βρυξελών ενώ αυτό απαγορεύεται και το έχω καταγγείλει επανειλημμένα σε αυτή την αίθουσα και έχω ζητήσει εξηγήσεις από την Κομισιόν και δεν παίρνουμε καμία απάντηση και πάλι προημερών συνέβη το ίδιο επομένως το να θέλουμε να βάλουμε μια τάξη στο ποιοι έρχονται στα σύνορα και εν συνεχεία στην ευρωπαϊκή ένωση είναι σημαντικό αλλά το να επιτρέπεται επαναφορά παρανόμων ελέγχων από το βέλγιο την αυστρία και άλλες χώρες σε όσους ταξιδεύουν από την ελλάδα είναι απαράδεκτο. Thank you, um, Ευχαριστώ. Ε, που θα χαλάσω την ωραία ατμόσφαιρα για να σκάσω τη φούσκα της ε, αγάπης. Τα έθνη, τα σύνορα είναι αρμοδιότητα των εθνών κρατών, όχι ενός υπερκράτους. Και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα της υπερσυγκέντρωσης που βλάπτει τα επιμέρους έθνη κράτη. Οι άνθρωποι από την Ελλάδα είναι διαφορετικοί από αυτούς της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Διαφορετικοί είμαστε και ευτυχώς. Καλή τύχη λοιπόν σε όλους όσοι φεύγετε. Δυστυχώς πολλά από αυτά που κάνατε ήταν παραπλανημένα και, για... και αυτό είναι από τα... μια από τις χειρότερες ιδέες αυτού του κοινοβουλίου. Τι να κάνουμε, μια φορά φεύγει ο καθένας μας. Η κυρία Τόμασιτς. Πρόεδρε, η σημαντικότερη νέα διάταξη είναι να είναι το ότι μπορούμε να ελέγχουμε τι επανεισδοχέ. Καλωσορίζω λοιπόν τη δημιουργία ενό μηχανισμού που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί την πολιτική θεωρήσεων για να παροτρύνει τις τρίτες χώρες να συνεργάζονται στα θέματα επανεισδοχής. Επίσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το ότι η πολιτική θεωρήσεων σχετίζεται με το πόσο Φιλικέ στην επανεισδοχή είναι τα κράτη. Μπράβο, επιτέλους το κατάλαβε. Ελπίζω ότι στη νέα Επιτροπή και στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αλλάξουν βασικά κομμάτια της πολιτικής θεωρήσεων. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα ζητήσω τώρα από τον Επίτροπο κύριο Κανιέτε να λάβει το λόγο. Ας τον ακούσουμε. Πρόεδρε, αξιότιμη, βουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική αυτή συζήτηση. Το νέο κανονισμό θα εξεχρονίσει την κοινή πολιτική για τι θεωρήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να διευκολυνθεί η πρόσβαση, για να είναι ίση η πρόσβαση για όλου του ετούντε και να προωθηθεί το ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για επιχειρήσει και για αναψυχή. Να είναι ίση η μεταχείριση όλων αυτών που ταξιδεύουν για τουριστικούς σκοπούς και για επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και πολιτισμική ανταλλαγή και πέραν αυτών οι νέοι κανόνε θα βελτιώσουν τη δυνατότητά μα να αντιδράσουμε και να δώσουμε, θα μας δώσουν ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για τη συνεργασία με χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τι επιστροφέ παρανομών μεταναστών. Ελπίζω να υποστηρίξετε τον συμβιβασμό σε ό,τι αφορά το νέο κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θεωρήσεις. Θα σας εξασφαλίσω και θα την βεβαιώ από πλευράς μας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδραματίσει το ρόλο που χρειάζεται για την εφαρμογή των αυτών διατάξεων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επιτροπέ Κανίτελα και ο Πρόεδρος, ο συνάδελφος Λόπες Αγγιλάρα. Έχει τώρα το λόγο. Ε, ήταν πολύ επικοδομητική η πλειοψηφία των παρεμβάσεων και αυτό δείχνει ότι μάλλον θα ψηφίσουμε υπέρ. Γνωρίζω ότι αυτό Τότε το κοινό νομοθέτημα θα δώσει απάντηση σε, αυτούς τους, ε, σε αυτά τα 70, 80, 90 εκατομμύρια άτομα που ε, επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νόμιμα κάθε χρόνο και προέρχονται από περισσότερες από 150 χώρες. Η δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τελειώνει ποτέ, οπότε σαφέστατα έχουμε πολλές εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, να δώσουμε απάντηση στο ανθρωπιστικά Τίματα ατόμων τα οποία ε, προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διοκόμενα, καταδιοκόμενα στη χώρα τους και δεν μπορούν να έρθουν νομίμως ε, εκθέτοντας την ε, ζωή τους σε κινδύνους για την ακαιρεότητά τους ή πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απαντήσει στο αίτημά μας το οποίο έχει γίνει, έχει υποβληθεί. Στην επόμενη θητεία λοιπόν θα πρέπει να υποβάλει μια πρόταση για ένα σύστημα ανθρωπιστικών θεωρήσεων, μια νόμιμη οδό προκειμένου αυτά τα άτομα, τα απελπισμένα άτομα που φεύγουν, προσπαθούν να ξεφύγουν από τι διώξει να φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νόμιμο τρόπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα είδου τέτοιο νόμιμο τρόπο χωρί να εκτεθούν και να εκθέσουν τη ζωή του και την ακεραιότητά του σε κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ όλου και όλε για τη συνεισφορά σα. Συνάδελφοι, ευχαριστώ που ήρθατε τόσο πολύ για να δω πώς σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γιατί και εγώ τελευταία φορά παρεμβαίνω με επίσημη ε, θέση στο, στην Ολομέλεια. Καλή επιτυχία και καλή τύχη σε όλους σας. je vous monsieur je suis Χαίρομαι που σας βλέπω να προεδρεύετε την τελευταία συνεδρίαση ψηφοφοριών εδώ στο Κοινοβούλιο. Α, όχι, όχι, έχει και αύριο, έχουμε και αύριο, έχουμε και αύριο, συγγνώμη. Θα είμαι εδώ. Μην ανησυχείτε, ηρεμήστε. Ξέχασα την αυριανή συνεδρία ψηφοφορία. Δεν υπάρχει περίπτωση να το σκάσω, να κάνω κοπάνα. Μία φορά νομίζω έχω κάνει κοπάνα. Ε, όταν ε, έκανα χείριση στην πλάτη. Αν μου επιτρέπετε να απευθύνω στον κύριο Κανιέτε που είναι εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Εδώ και κάποιους μήνες το Κοινοβούλιο ανέφερε στην ε, Κομισιόν, που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, ότι υπάρχει μια ενδεχόμενη κατάσταση σύγκρουση συμφερόντων σε ό,τι αφορά έναν Πρωθυπουργό της Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτόν της Τσεχίας. Τη Δευτέρα μα πέρασε ο Επίτροπο Έτιγκερ, εμφανίστηκε στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τι μα είπε. Μα είπε ότι πράγματι υφίσταται τέτοιου είδου περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων, αλλά θα πρέπει να το μελετήσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν είμαστε σίγουροι, πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μα κλπ. Διαπιστώνουμε <clears throat> ότι οι αστυνομικέ αρχέ τη Τσεχία ε, κατηγορούν προσωπικά τον Πρωθυπουργό της Τσεχίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα αναρωτιέται. Τι να καταλάβω από αυτό κύριε Κανιέτε, ότι η Κομισιόν έχει πολιτικό κίνητρο να αναβάλει την εργασία της ε, παραμελώντας το ρόλο της ως ε, θεματοφύλακα των συνθήκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν μπορεί να προχωρήσει αν υποψιαζόμαστε ότι κάποιοι ηγέτες μας πλουτίζουν παράνομα. Γι' αυτό το λόγο εσείς θα πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Merci, Le de vous était Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Λαμπέρ και ελπίζω ότι θα σας ξανακούσουμε. Κύριος Βιώτη. Σας ακούμε, ακούμε τον κύριο Βιώτη κύριε και κύριοι. Παρεμβαίνω πρόεδρε, διότι βρίσκω απαράδεκτο να μην συζητάμε στο σώμα αυτό ούτε με μια λέξη για το τι γίνεται στη Λιβύη, όχι τον πόλεμο, αλλά αυτό που υφίστανται 200.000 περίπου πρόσφυγες που εγκαταλείπονται εκεί να πεθάνουν στα, στρατόπεδα συγκέντρωσης, που θα εξαφανιστούν από τις βόμβες ενός ε, πολέμου που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ας ζητήσουμε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ξανανοίξουν τους δρόμους για τις ΜΚΟ, να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Ας ζητήσουμε από τις, ε, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να απελευθερώσουν τον δρόμο και να ξαναφέρουν στην Ευρώπη, αυτά τα γυναικόπαιδα που βρίσκονται στον πόλεμο. Αυτό είναι ο ρόλο του Κοινοβουλίου, αυτό είναι ο ρόλο μας. Ευχαριστώ κύριε Βιώτη. Συνάδελφοι, λίγη ησυχία. Ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό χρειάζομαι και δεν θα λυπηθείτε. Και νομίζω ότι είναι πρόκληση για τους διερμηνείς. Έψαξα να βρω, αλλά δεν είδα την παράγραφο που έχετε υπόψη για μια τελευταία ε, παρέμβαση εδώ πριν καθαρίσει ο χρόνος ό,τι έχουμε κάνει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ευχαριστώ όχι προς τους πολλούς φίλους, άντρες ή γυναίκες, αλλά και σε όσους εργάζονται εδώ, στο μπαρ που μας δίνουν μπύρες, που ε, διανέμουν τη λίστα ψηφοφορίες, ε, που είναι στο γκαράζ, στη... μας δίνουν αυτοκίνητα, τόσους πολλούς ε, που τους έλεγε σε πολλές γλώσσες προχωρήστε, σταμάτα, κάτσε λίγο, πήγαινε πιο γρήγορα. Αυτούς που μας έδιναν τα μπάτζ που ήταν πάντα ευγενικοί. Και θέλω αυτούς που μεταφράζουν τους, ε, τις ομιλίες και που παλεύουν τώρα με αυτά που λέω. Θα τελειώσω όμως τώρα και μετά θα αλλάξω καιρός. Ευχαριστώ λοιπόν σε όλους. Ευχαριστούμε κύριε Φρόιντ. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα τι ομοιοκαταληξίε σα και τι αξιολόγησα όπω θα έπρεπε, αλλά περνάμε στι πληροφορίε. Έκθεση. Κυρία Μιράντα. Παρακαλώ. Ε, τώρα που τελειώνουμε τη θητεία μας, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 7 του κανονισμού, να το επικαλεστώ για να δούμε λίγο την κατάσταση δύο πρώην ευρωβουλευτών των πράσινων. Πάνω από 500 μέρες βρίσκονται στη φυλακή. Ραούλ Ρομέβα Ιρουέβα και Ουριόλ Χιουνκέρας. Αυτά είναι τα ονόματά τους. Αυτός ο τελευταίος είναι επικεφαλής υποψήφιος ε, για, τις, ε, ε, για την ελεύθερη συμμαχία της Ευρώπης. Et enfin, Κύριο Κούλογλου, κύριε Κούλογλου, παρακαλώ να είστε σύντομο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ήθελα να σα ε, ζητήσω τη βοήθειά σα και να ζητήσω και τη βοήθεια των συναδέλφων. Ήμουν μέλο μια επίσημη αντιπροσωπεία ε, δι δύο φορέ ε, στι ΗΠΑ, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και μου αρνήθηκαν τη χορήγηση θεώρηση και να μπω στι ΗΠΑ. Με μισό λεπτό, μισό λεπτό περιμένετε. Περιμένετε, παρακαλώ δεν έχω να κάνω τίποτα με την τρομοκρατία. Επειδή είμαι δημοσιογράφος, παραγωγός των ιών, ξέρω ότι με τον Τραμπ είσαστε εσείς, μην ανησυχείτε, το ξέρω. Ξέρω από πού είσαστε. Κύριε Κούλογλου, λέει η πρόεδρος, παρακαλώ παρουσιάστε το σημείο σας. Απέστειλα επιστολή προς τον πρόεδρο Ταγιάννη, δεν έλαβα απάντηση. Αναζητώ λοιπόν και ζητώ τη δική σας βοήθεια και τη βοήθεια όλων των δημοκρατών συναδέλφων. Όχι εσάς, εσάς δεν κάνετε βοήθεια σας της άκρας δεξιάς. Μάλιστα κύριε Κούλογλου, ε, μάλιστα κύριε ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Euh, Περνάμε στις ψηφοφορίες με την έκθεση Σάγερ. Ενία ψηφοφορία, μια μοναδική ψηφοφορία, ονομαστική, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Κλείνουμε την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Δεύτερη έκθεση του κ. Σάγερ. Ονομαστική ψηφοφορία για την, ε, για την τροπολογία 585. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 586. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 587 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Κλείνει η πρώτη ανάγνωση. Τρίτη έκθεση Σάγερ. Μοναδική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου άρχεται. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κλείνει η πρώτη ανάγνωση. Περνάμε στην έκθεση Αρτουή. Κύριε Αρτουή, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ, είναι συντομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η τελευταία μου παρέμβαση στην Ολομέλεια. Η έκθεση που υποβάλλω προς ψηφοφορία, προς ψήφιση, ε, είναι ε, ένας ε, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει σκοπό να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Ένα προπολογισμό πολύ μικρός, 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ και αυτός εξαρτάται από τις ε, εθνικές συνσφορές. Ε, θα ήθελα, φεύγοντα από εδώ, να συμμεριστώ μαζί σας καταρχήν το, ιδανικό, το, το όραμά μου. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια παγκόσμια δύναμη. Ο φόβο μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πολύ διατεθειμένα να αυξήσουν τι συνεισφορές τους. Και η πεποίθησή μου είναι ότι η αύξηση του προπολογισμού, του ευρωπαϊκού προπολογισμού, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ελάφρυνση των εθνικών προπολογισμών. Αυτό θα σήμαινε μεταφορέ κονδυλίων από του εθνικού προπολογισμού στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οπότε η επιθυμία μου και η ευχή μου είναι στην επόμενη θητεία να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα αυτός ο κοινό ευρωπαϊκός παρανομαστής ε, που εξαιτία της παγκοσμιοποίησης τα κράτη-μέλη σε εθνικό αποκλειστικά επίπεδο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στο μέλλον. Χαιρετίζω την προσήλωσή σας, συνάδελφοι, και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμού. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάχημη καθημερινά, θα ήθελα ε, να πω ότι αυτό οφείλεται σε εσά και σε μας. Ε, τα, την ευγνωμοσύνη μου. Ζήτω Ευρώπη, ζήτω τα κράτη-μέλη. Ψηφίζουμε την έκθεση Αρτουή. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Έκθεση Eller. Νόμο ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Χούμπνερ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του κανονισμού εγκατάσταση και λειτουργική χρήση συνεργατικών εφιών συστημάτων μεταφορών. Ψηφίζουμε επί του ψηφίσμα στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα το επιβεβαιώσουμε, θα το επαληθεύσουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ψήφιση της έκθεσης Μέτσολα. Ε, πρόταση απόρριψης πρόταση Κομισιόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε στην στην, τροπολογία, στην ψήφιση τροπολογίας 5-12 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 513 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίγη η πρώτη ανάγνωση από του Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Λόπες Αγγιλάρ. Που θα ήθελα να πάρει το λόγο αν καταλαβαίνω καλά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ένα λεπτό κι εγώ. Είναι η τελευταία ψηφοφορία για ένα σημαντικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τον κώδικα θεωρήσεων. Και ήθιστε πριν την ψηφοφορία στην Ορομέλεια και ενώπιον όλων των μελών να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την επικοδομητική συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους κοιόδης συζητητές στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, τον πρόεδρο και συνάδελφο Κλοντ Μωράες. Αλλά με δεδομένο ότι αυτή είναι η τελευταία ολομέλεια του Κοινοβουλίου μας, καλό θα ήταν να, και σύνθεση είναι να εκφράσουμε δημοσία την η ικανοποίησή μου που μπορέσαμε να υπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες στο σώμα αυτό, το μόνο ερετό δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα αυτής της του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και να σας ευχηθώ πραγματικά εκ βάθους καρδίας ό,τι καλύτερο για όλους και να σας πω ότι είναι, ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σας τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευχαριστώ όλους σας συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε και εμείς κύριε Λόπες Αγγιλάρ. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πρώτη ανάγνωση ολοκληρώνεται. Έκθεση Σεράο Σάντο. Και εδώ ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 82. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται. Προχωρούμε. Έκθεση Ράντεφ. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 73 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Ψηφοφορία για την έκθεση Ρέντα. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρούται έτσι. Έκθεση Βίρκουνεν Μαρινέσκου και Τελιτσκα. Τροπολογία 108 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές, θα γίνει έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρόταση με ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο της Επιτροπής. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται. Έκθεση Ντάλτον. Τελειώνουμε με αυτήν. Τροπο, πολλές τροπολογίες της, Επιτροπή, της αρμόδιας Επιτροπής ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία η τροπολογία 31 άρχεται η ψηφοφορία. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο για το 19. Ωραία. Έλεγχος για το, την τοπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. 19. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία η τροπολογία 31 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 59 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές, δεκτή. Με ονομαστική ψηφοφορία 63 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67 άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία πάλι. Πέρας. Δεκτή. 82 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 87. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ονομαστική ψηφοφορία για το 163 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 66 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Έλεγχος για την 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 160. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Η 66 υπερψηφίστηκε, άρα πηγαίνουμε στην 160. Ψηφίζουμε την 160 με ονομαστική ψηφοφορία. Πάντα ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 157. Άρχεται η ψηφοφορία. 157. Πέρας. Απορρίπτεται. 164. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 81. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η επόμενη. 83D με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Προχωρούμε λοιπόν στην 85. Όλες οι άλλες καταπίπτουν. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι σίγουρη. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Να σηκώνετε το χέρι σας αν γίνεται. 86. Γιατί όλες οι υπόλοιπες, η 175 πέφτει. 86 δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Λυπάμαι αλλά δεν σηκώνονται τα χέρια σας. Θα γίνει λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 86D, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 88. Γιατί έχουν καταπέσει οι προηγούμενες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 165 Δε. Ναι, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Με ονομαστική ψηφοφορία 161. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 162. Άρχεται πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Με ονομαστική ψηφοφορία 158. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και 156 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε Δε. υπέρ, κατά, αποχές θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 18η άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 159. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορια περας ψηφοφοριας Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές. Ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται και ολοκληρώνεται.